Καλώς ήλθατε στο πρώτο αυτό μέρος της συνεδριάσεως. Πρόκειται για ενημέρωση, debriefing δηλαδή, για τις εκλογές στην Μολδαβία που έλαβαν χώρα στις 30 Νοεμβρίου και στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας τους αποδίδουμε στις εκλογές δηλαδή μεγάλη σημασία. Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις πέτυχαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχουν μπει τώρα σε δύσκολες συζητήσεις για τη δημιουργία συνασπισμού. Ελπίζω ότι οι συζητήσεις αυτές θα διεξαχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι εσωτερικές συγκρούσεις. Να μην χαθούν δηλαδή οι πραγματικές ανάγκες από τα μάτια γιατί καμιά φορά τυχαίνει να χάνει τις εκλογές κανείς μετά, στις εβδομάδες που ακολουθούν. Ελπίζω λοιπόν ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ιδίως στην Πολωνία, λέει κάποιος χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, είχαμε και αποστολή εκεί με συνδυασμό σε συνδυασμό με τον ΟΑΣΕ και Επίσης, ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την διεύθυνση του Σόλτες. Ελπίζω θα μπορέσει να μας εξηγήσει τι έγινε. Χαίρομαι. Μπορέσαμε, κάνουμε την ενημέρωση αυτή σε συνδυασμό, σε συνεργασία μάλλον με την ε, κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία και ευτυχώς είναι και παρόν ο κ. Κριστέα. Πριν να δώσω τον λόγο στον κύριο Σόλτης. Κύριε Κριστέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε ήδη σωστά ότι οι εκλογές στην Δημοκρατία της Μολδαβίας έχουν μεγάλη σημασία. Ίσως είναι πλέον σημαντικές από τότε που κηρύχθηκε αυτή η χώρα ανεξάρτητη. Δεν θέλω να προχωρήσω ευθύ αμέσω στα συμπεράσματα των ε, αποστολών παρατηρήσεων εκλογών. Ο κύριος Ευωζόλτες θα το πράξει αυτό. Εγώ ήθελα να πω εν προκειμένου ότι συνεργαστήκαμε καλά. Η αντιπροσωπεία εμφανίστηκε ενωμένη και στην τελική έκθεση πέρασαν τα μηνύματα που θέλαμε εμείς στην τελική έκθεση των τριών διεθνών οργανισμών που άσκησαν την παρατήρηση των εκλογών. Δυστυχώ. η προεκλογική εκστρατεία εμφανίστηκε πολύ πολλωμένη. Ο προεκλογικό αγώνας στην Δημοκρατία της Μολδαβίας διαρκεί 60 ημέρες. Εκεί, όπως είπα, η ατμόσφαιρα ήταν έντονα φορτισμένη συναισθηματικά οι εκλογές είχαν και γεωπολιτικό χαρακτήρα περισσότερο και λιγότερο κοινωνικο-οικονομικό χαρακτήρα, ας το πω έτσι. Τους απασχόλησε πολύ η κατεύθυνση της χώρας τους. Προτεραιότητα υπαριθμών ένα θα είναι τώρα η Συμφωνία Συνδέσεως για την κυβέρνηση που θα δημιουργηθεί. Ήδη έχουν ψηφιστεί ορισμένοι νόμοι αλλά είναι πολύ σημαντικό τώρα όλοι αυτοί να μπορέσουν να εφαρμοστούν, ιδίω για να επιτύχει η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, δεν είναι ακόμα σαφές αν θα μπορέσουν να γίνουν. Η νέα κυβέρνηση ελπίζουμε ότι θα είναι η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση που αναμένουμε και ελπίζουμε ότι θα επιτύχει να δράσει με τρόπο αποτελεσματικό, διότι ο χρόνος πιέζει. Και αυτά τα είπαμε και επί τόπου, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους εκεί. Επίσης σημαντική είναι η διατήρηση της συνέχειας. Πρέπει να αποφευθεί παραπέρα πόλωση της κοινωνίας. Πρέπει να ενταχθούν οι μειοψηφίες στον κοινωνικό διάλογο για να μειωθούν οι εντάσεις. Κάτι που είναι σημαντικό είναι και εμείς από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωση, να πιέσουμε αλλά και να υποστηρίξουμε. Πρέπει να ταχθούμε στο πλευρό τους και να τους συνοδεύσουμε στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Αυτό το θέλουν οι πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Αυτό ψήφισαν στις 30 Νοεμβρίου. Ψήφισαν μια φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία. Και μάλιστα στο κοινοβούλιο τους έχουν εξασφαλίσει πλέον επαρκή πλειοψηφία. Ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον κύριο Μαουρίτσιο Μάκρη δήμαρχο, αρχιδήμαρχο του Μπουένος Άιρες. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις εργασίες μας και σας διαβεβαιώ ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη χώρα σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τον Μέρκοσούρ προς το συμφέρον αμφωτέρων των πλευρών. Σας ευχαριστώ και πάλι που διαθέτετε αυτόν τον χρόνο για να παρακολουθείτε τις εργασίες μας. Das Wort Κύριε Σόλτες. Σας ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σας μιλήσω ως επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Διεθνή Επιτροπή Παρατήρηση Εκλογών ε, στη Μολδαβία. Ήμασταν λοιπόν, όπως είπα, μέλος ε, της ε, διεθνούς αντιπροσωπείας και ως Κοινοβούλιο συμφωνούμε με τα προκαταρκτικά απορίσματα και συμπεράσματα της έκθεσης της αποστολής παρατήρησης και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν επίσης στην αποστολή αλλά και τους συναδέλφους ε, άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων και επιτροπών και θα ήθελα να πω ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Η ομάδα μας παρατήρησε τις εκλογές ε, στα διάφορα τμήματα της χώρας, σε διάφορα εκλογικά τμήματα. Επισκεφθήκαμε λοιπόν ε, πολλά ε, εκλογικά τμήματα, μεταξύ αυτών και κάποια συγκεκριμένα, παραδείγματος χάρη διοικητική γραμμή με την υπερτινιστερία όπου τα, οι κάτοικοι της περιοχής αυτής μπορούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα ε, ψήφου που δεν μπορούσαν να ασκήσουν στις περιοχές που κατοικούν, που διαμένουν. Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από μια ε, ευρεία επιλογή, ε, υπήρχαν πολλές επιλογές, διοικητικά πήγαν καλά επίσης. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση, μεγαλύτερη τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές παρότι είχε υποθεί ότι υπήρχε μια γενική απάθεια και έλλειψη ενδιαφέροντος και υπήρξε μια άνετη πλειοψηφία των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων. 55 έδρες, σοσιαλιστές κομμουνιστές 46 έδρες μαζί. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή είχε απαγορεύσει το κόμμα Πάτρια γιατί ε, είχε δεχθεί παράνομη χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Οι ψηφοφόροι λοιπόν άσκησαν το δημοκρατικό τους δικαίωμα με ειρηνικό τρόπο, ε, με ομαλότητα, χωρίς να υπάρχουν ε, προβλήματα και παρατυπίες, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό. Ήταν υψηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων στις περιοχές που επισκεφθήκαμε. Ψήφισαν ελεύθερα οι Μολδαβοί, και το νεοεκλεγέν κοινοβούλιο θα πρέπει άμεσα να αρχίσει να υλοποιεί τις ε, εδώ και καιρό αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις ε, για ε, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα, καταπολέμηση της διαφθοράς, τη χρηματοδότηση των κομμάτων, εκλογικός νόμος, είναι μερικά από τα θέματα. Υπήρχαν σημαντικές προκλήσεις για τις εκλογές λόγω και της ε, γεωπολιτικής θέσης και αυτά κυριάρχησαν και στην προεκλογική εκστρατεία. Τα κοινωνικά οικονομικά ζητήματα ίσως τέθησαν σε δεύτερη μοίρα. Υπήρξε πόλωση της κοινωνίας. Πάντως οι ψηφοφόροι ε, έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στις εκλογές. Η χώρα τώρα πρέπει να αντιλήσει το δυναμικό αυτό, να το εκμεταλλευτεί τα μάλα. Σημειώσαμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στη χώρα. Είδαμε όμως ότι υπάρχουν και ακόμη κάποιες αδυναμίες, κάποιες ελλείψεις. Τονίζουμε ιδίως την ανάγκη η σύσταση της αποστολής παρατήρησης ε, του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΑΣΕ, ο και θέλουμε επίσης να επιμείνουμε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ελευθεροτυπίας και της πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωση. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης διαφάνεια και στην ιδιοκτησία των μέσων επικοινωνίας. Ως τελευταίο σημείο να πω ότι ναι μεν χαιρετίζουμε και την ε, υψηλή εκπροσώπηση γυναικών στα διάφορα εκλογικά τμήματα, αλλά θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να ε, υιοθετήσει τα νομοσχέδια ε, που ήδη είναι υποσυζήτηση για μεγάλη, μεγαλύτερη ε, συμμετοχή των γυναικών που παραμένει χαμηλή, ιδίως σε κάποιες ευάλωτες θέσεις. Και βέβαια όλες οι ε, μειονότητε, θα πρέπει τα δικαιώματά του να γίνουν σεβαστά μεταξύ αυτών και των Ρωμά. Επαναλαμβάνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με το νέο Μολδαβικό Κοινοβούλιο ε, περιμένει την συνεργασία μας στο πλαίσιο της κοινοβουλευτική Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Θα πρέπει η όθηση να παραμείνει ε, σε αυτό το επίπεδο για την υιοθέτηση φιλόδοξων πολιτικών που θα ωφελήσουν όλους τους Μολδαβούς. Πιστεύω ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν άλλη ευκαιρία πρέπει πλέον να γίνει πραγματικά στροφή 180 μοιρών. Και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει και αυτή μια αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και την ομαλή εφαρμογή της νέας συμφωνίας τερικής σχέσης, που σίγουρα δεν είναι και ο απότατος στόχος των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Είναι απλά ένα κομμάτι ε, της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που καταβάλατε αυτή την προσπάθεια και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας σας ε, αυτής της αποστολής. Η κυρία Καλνιέτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στη Μολδαβία εμείς Τρία μέλη, δηλαδή εγώ, ο κύριος Γκάλαρ και ο κύριος Τσέτινα, επισκεφτήκαμε τη χώρα και συμμετείχαμε και σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Το μήνυμα που εμείς διαβιβάσαμε εκεί είναι ότι τώρα υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη, αλλά μετά από τις εκλογές ε, μπορεί κάπως να χαλάσουν οι σχέσεις μας. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν ε, μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικοί που είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων να καταλάβουν ότι αυτές είναι πήγουσες. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει πάρα πολύ συγκεκριμένα να εκπονήσει έναν οδικό χάρτη που να βασίζεται στη συμφωνία σύνδεσης και θα βοηθήσει τους πολιτικούς, θα τους πλαισιώσει για όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν. Και θα πρότεινα το εξής δεν θα μπορούσαμε να συστήσουμε ομάδες εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένα καθήκοντα. Ας πούμε κάποιες τέτοιες task, task forces, ομάδες εμπειρογνωμόνων που να υποβοηθούν. Συνήθως τέτοιες ομάδες απαρτίζονται από ειδικού εμπειρογνώμονες από χώρες της προανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικές γιατί είναι χώρες στις οποίες ε, κυριαρχούσε η Σοβιετική Ένωση και χρειάζεται πολύ μεγάλος μετασχηματισμός και μεταρρύθμιση. Θα πρέπει η Μολδαβία λοιπόν να ε, χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές και να μάθει και από τα λάθη τους, γιατί είναι η ίδια διαδικασία μετασχηματισμού. Και ε, ε, η νεεκλογήσα τώρα κυβέρνηση θα πρέπει να προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα που είναι βαθύ στη Μολδαβία. Εάν δεν είναι σε θέση τώρα, σε αυτή τη μεταγλογική περίοδο, να πείσουν ότι τουλάχιστον 20% του πληθυσμού ε, παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίξει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τότε υπάρχει κίνδυνος οπισθοδρόμησης ε, στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή δεν έχει αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος, εξακολουθεί να ισχύει. Ευχαριστώ. Um... Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Donc, euh, pour... Λοιπόν, δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Γι' αυτό άλλωστε ζήτησα και το λόγο. Έγιναν εκλογές στη Μολδαβία, πήγαν καλά. Εγώ θεωρώ απολύτως γελίες τις κριτικές για την απαγόρευση ενός κόμματος. και τον αποκλεισμό του από την εκλογική αναμέτρηση, διότι απλούστατα επρόκειτο για την απαγόρευση ε, ε, να μπει στο ε, προεκλογικό αγώνα ένα κόμμα που είχε παράνομη χρηματοδότηση, προκειμένου από τη Μόσχα. Δηλαδή, εμείς επικρίνουμε τη Μόσχα και τα ευρωπαϊκά δημοσιεύματα και κάποιες πολιτικές ομάδες. Και αν συμμετείχε αυτό το κόμμα θα προσανατόλιζε από την πραγματική εκλογική αναμέτρηση και από το διακύβευμα, γιατί επρόκειτο ακριβώς για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Μολδαβίας και το εκλογικό σώμα το υπερψήφισε. Οποιαδήποτε διαφορετική ανάγνωση ε, παραγνωρίζει την ουσία. Ένα ε, δεύτερο που ήθελα να πω είναι το εξής. Απομένουν πολλά ακόμα να γίνουν σε δύο τομείς και ελπίζω ο κυβερνητικός συνασπισμός που είναι τώρα υπό σχηματισμό ε, θα το κάνει προτεραιότητες. Λοιπόν, πρώτον, θα πρέπει γρήγορα να γίνουν πρόοδοι. Είναι να ε, τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα το καυτό πρόβλημα. Η ε, δημοκρατία της Μολδαβίας δεν πρόκειται να προχωρήσει εάν δεν, να το πω, τροποποιήσει σαφέστατα τη στάση της σε σχέση με αυτό. Πολύ δε περισσότερο ε, που ε, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν δουλειά οι Μολδαβοί αλλού. Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να παταχθεί η ε, διαφθορά. Είναι απολύτως απαράδεκτα αυτά να αναβάλλονται. Είναι δύο ταυτόχρονες λοιπόν προτεραιότητες. Δουλειές να δημιουργηθούν και να παταχθεί η διαφθορά. Οπωσδήποτε. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ξεκάθαρα και εκεί θα κριθεί τελικά και η κυβέρνηση. Ανάλογα με τη στάση της ως προς αυτό. Τέλος θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μετέβησαν εκεί για την παρατήρηση των εκλογών. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Colleagues, uh, in fact, uh, the results in Moldova Αγαπητοί συνάδελφοι, τα αποτελέσματα της Μολδαβίας ε, ε, είναι απόδειξη ότι πολύ καλά ε, τον Οκτώβριο χειριστήκαμε την κατάσταση με την έγκριση της Συμφωνίας Σύνδεσης. Είναι επιβεβαίωση λοιπόν της πορείας που έχει πάρει η χώρα, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι πολύ σωστά. Στη διάρκεια των εκλογών υπήρχε μια γραμμή πόλωσης ε, μεταξύ Βρυξελών και Μόσχας κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε άκρος ε, λαϊκιστικές ε, δηλώσεις από κάποιους σοσιαλιστές πολιτικούς στη Μολδαβία, οι οποίοι μάλιστα χρησιμοποίησαν αφήσεις του εαυτού τους με τον Πούτιν, πολύ απλά για να δείξουν ότι με αυτόν συντάσσονται. σαν να μην έχει η χώρα καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συμφωνία Σύνδεση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η τακτική τη πόλωση, αλλά αυτό πρέπει όλοι μα να το δούμε ω ένα κίνητρο για να μην αφήσουμε μόνη τη τη Μολδαβία μετά από αυτέ τι εκλογέ. Αντιθέτω, πρέπει να συνεχίσουμε την συνεργασία μα και την παροχή βοήθεια ε, σύμφωνα με τι διατάξει του όρου τη Συμφωνία Σύνδεση. Βλέπουμε όμως ο πληθυσμός ε, να κοιτάει και προς τα πίσω, προς το παρελθόν ακόμη. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βελτιώσουμε και την ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τι δυνατότητες ε, έχει και προσφέρει αυτή η συμφωνία σύνδεσης και πιστεύω ότι ο συνάδελφος Αντικριστέα θα κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε θα υπάρξουν περισσότερες επαφές ε, με ευρωβουλευτές από τα ταξιδέψουν στη Μολδαβία και θα συνομιλήσουν με τον κόσμο εκεί για να ενημερώσουν ε, το λαό της χώρας. Επίσης ε, φυσικά και πρέπει να συγχαρούμε τη Μολδαβία. 55-46 το αποτέλεσμα δεν φαίνεται ίσως τόσο σταθερό εντό αγωγικών, αλλά είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Δεν εκρίθηκε με μια ψήφο διαφορά, ε, η εκλογική αναμέτρηση. Σίγουρα ε, τα δύο μπλοκ έχουν μία διαφορά και ελπίζω το φιλοευρωπαϊκό μπλοκ να κυβερνήσει με σταθερότητα και να μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Thank you, um, ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, μια απαγόρευση κομμάτων από τις εκλογές επειδή χρηματοδοτούνται από τη Ρωσία. Αν γίνει αυτό ρουτίνα πλέον στην Ευρώπη, πιστεύω ότι ορισμένοι συνάδελφοι θα ανακουφιστούν από κάποιες μεγάλες ανησυχίες που τρέφουν. Όχι, εντάξει, αστείευομαι. Αλλά θέλω να πω ότι προσωπικά αυτό το αποτέλεσμα δεν μου φαίνεται και τόσο λαμπρό ή σπουδαίο, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι και το περιέγραψαν. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είναι πάρα πολύ γερή, αλλά αυτή δεν υποστηρίζεται από λαϊκή βάση ε, πλειοψηφία. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια κόμματα που δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή και, ε, γιατί δεν πέρασαν το κατόφλι. Και αν ε, υπολογιστούν και αυτά νομίζω ότι βαδίζει σε κάπως αβέβαιο και σαθρό έδαφος η κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε μαζί τους έτσι ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αυτή πορεία και ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός τους. Για να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να απευθυνθούμε και σε εκείνους που είναι στην άλλη πλευρά για να μπορέσουμε να τους κερδίσουμε υπέρ της Ευρώπης και ενδεχομένως να χρειαστεί και ιδιαίτερη προσπάθεια. Και ίσως να πρέπει να συζητήσουμε και με κάποιες άλλες δυτικές δυνάμεις για τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της Μολδαβίας. Δεν είμαι πάντα βέβαιος ότι οι Αμερικανοί το βλέπουν από την ίδια σκοπιά με εμά αυτό το θέμα. Μήπως να το συζητούσαμε και μαζί τους, γιατί και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τον επίγοντα χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων και την ενδιαφέρουσα πρόταση που κατέθεσε η κυρία Καλνιέτε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής οι κυβερνήσεις των χωρών το προτείνουν. Αναφερθήκατε σε κάποιε χώρε, υπενηχθήκατε κάποιε χώρε. Ποιο θα δώσει αυτή τη βοήθεια, οι κυβερνήσει ή η κοινωνία των πολιτών. Έχουν εκφράσει προθυμία και από την άλλη η μολδαβική κυβέρνηση έχει εκφράσει προθυμία να δεχτεί τέτοια βοήθεια. Και από πλευρά θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχει και πάλι προθυμία να οργανώσει όλη αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσει και να υποστηρίξει τη μολδαβική κυβέρνηση. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που ασχολούνται με αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε και τη διαδικασία επιγόντως ό,τι αφορά τις δικές μας συνεισφορές και δράσεις. Γιατί είναι, είναι τώρα ευκαιρία, αλλά είναι μικρή και στενή χρονικά η ευκαιρία. Oh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτό απατώμεθα, αυτό το άθλημα εξασκούμε αυτή τη στιγμή. Α, δεν ήταν η σειρά σα. Ήσασταν μέλο του ECR, δεν το ξέρα, λέει ο πρόεδρο. you, Kippy? Yeah, yeah, yeah, yeah, Mr. Tan, look quite worried for a minute then. Thank you, Chair. It's been claimed here that pro-European Union parties won the Moldovan elections. How... Είναι σαφές ότι κέρδισαν τις εκλογές φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Υπάρχουν όμως ε, και κόμματα της αντιπολίτευσης ε, με μεγάλα ποσοστά, 20% και στην συνέλευση 25,6%. Και από το 2005 δεν είχαν γίνει, ε, στις εκλογές δεν είχαν πάρει πάνω από 5%. Προσπαθούν ε, τα ευρωπαϊκά κόμματα να πάρουν ε, ε, την πλειοψηφία στις εκλογές αυτές. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία που δεν ε, ταιριάζουν για το ποιος έχει και με, με ποια διαφορά ποσοστών την πλειοψηφία. Για να υπάρξει προσέγγιση Μολδαβίας, και Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να βασιστεί με κάποιο δημοψήφισμα. Τότε λοιπόν και καμία Βρετανική κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει ποτέ την πλειοψηφία αφού δεν ξεπερνάτε ποτέ το 37%. Ή μήπως δεν έχω κατανοήσει καλά το Βρετανικό σύστημα. Ο κύριος Τάνοκ, έχετε δίκιο. Δεν έχετε παρανοήσει. Ίσως κάποια στιγμή να κερδίσουν οι εργατικοί με 32-32% της λαϊκής ψήφου. Αυτό είναι μία από τις ιδιοσυγκρασίες του συστήματός μας. Πάντως, παρόλα αυτά, η Μαργαρίτα Θάτσερ είχε φτιάξει μια ισχυρή κυβέρνηση με 42 περίπου της εκατό της λαϊκής ψήφου. 45% της περισσότερες ε, δημοκρατίες που χρησιμοποιούν το πλειοψηφικό σύστημα είναι ένας υγιής αριθμός ψηφοφόρων. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ με τον κύριο Μπιουτικόφερ ότι δεν είναι και καμιά λαμπρή νίκη των προοδευτικών δυνάμεων που θέλουν να φέρουν τη Μολδαβία στην πορεία μιας ένταξης ε, στις ευρωατλαντικές σχέσεις και σε μια πιο φιλελεύθερη δημοκρατία. Στη χώρα μου δεν μπορώ να μιλήσω βέβαια για τον εσωτερικό νόμο της Μολδαβίας, πάντως ο Βρετανικός νόμος απαγορεύει οποιαδήποτε χρηματοδότηση από ξένες κυβερνήσεις κομμάτων, ακόμα και πολιτών. Επομένως όντως με ανησυχούν προσπάθειες ορισμένων κυβερνήσεων και ιδίως της Ρωσικής να προσεγγίσουν υπερβολικά ορισμένα πολιτικά κόμματα. Έχουμε σοσιαλιστές σε χώρες όπως Βουλγαρία και Μολδαβία Έχουμε όμως και την άκρα δεξιά, το ε, εθνικό μέτωπο στη Γαλλία, το οποίο λαμβάνει δάνειο από ρωσική τράπεζα. Αυτό είναι το ε, παράξενο παιχνίδι που παίζει η Ρωσία. Άλλωστε ο Winston Churchill είχε πει πλειοψηφία ενός μου αρκεί για να κυβερνήσω τη χώρα. Είναι μικρή λοιπόν η πλειοψηφία, ούτε είναι ιδιαίτερα στέρεα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη Μολδαβία και να της προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια για να στηρίξουμε την κυβέρνηση αυτή που είναι σαφώς εύθραυστη και για να εξασφαλίσουμε ώστε οι Μολδαβοί να κατανοήσουν ποια είναι τα ωφέλη από μια προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Αν θέλουν να επιστρέψουν στη Σοβιετική Ένωση, ε, θα χρειαστεί να πληρώσουν βαρύτατο τίμημα και με την προσωπική τους ελευθερία, αλλά και με την δημοκρατική τους ελευθερία. Δεν νομίζω ότι θα δυσαρεστούσε αυτό βέβαια τον πρόεδρο Πούτιν. Πρόκειται λοιπόν για μια ελαφρά απογοήτευση, ομολογώ, παρόλα αυτά να συνεχίσουμε να σκεπτόμαστε θετικά και να τίνουμε χείρα βοηθείας σε όλους τους Μολδαβούς φίλους μας και να τους ε, βεβαιώσουμε ότι είναι ευπρόσδεκτοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι επίσης ευρωπαϊκοί πόροι βοήθειας αλλά και εμπορικές παραχωρήσεις με βάση την Συμφωνία Συνδέσεως μπορούν να τους προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Και αν μπορέσουν να λύσουν και το πρόβλημα της υπερδνηστερίας, ακόμα καλύτερα. Φοβούμε ωστόσο ότι ο ίσως ο κύριος Πούτιν, τώρα που μιλούμε κιόλα, να λογαριάζει αν μπορεί να φτιάξει ένα διάδρομο μέσω της Μαριοπόλ στην Κρυμαία και να αρπάξει έδαφος λοιπόν και από τη χώρα αυτή. Ελπίζω αυτή η φόβη μου ωστόσο να μην αποδειχθούν αληθινοί. Τώρα ο κύριος Νάρτ. Bueno, ahora sí. Disculpe, señor presidente. Α, τώρα είναι η σειρά μου. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν είχα καταλάβει σε ποιον δώσατε το λόγο. Εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω με τα μαθηματικά και με τα ε, πραγματικά ε, γεγονότα. Δεν μιλώ για τι επιθυμίε μου ή τα ιδεώδη μου. Δεν κατανοώ λοιπόν γιατί έχετε κατενθουσιαστεί από τα αποτελέσματα των μολδαβικών εκλογών. Εγώ επιθυμώ να ενταχθεί η Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με βάση την πραγματικότητα και όχι τους ευσεβείς πόθους. Σοσιαλιστικό κόμμα που 601.000 ψήφοι που ήταν οι κομμουνιστές, φιλελεύθεροι δημοκράτες 710 ψήφοι. Χιλιάδες μάλλον. Ε, η χώρα είναι διχασμένη. Και βλέπετε εδώ πώς ε, κατανέμονται οι έδρες. Το κόκκινο είναι σοσιαλιστές και κομμουνιστές και το υπόλοιπο είναι εκείνοι που κέρδισαν. Είναι η χώρα ε, μοιρασμένη στα δύο. 55 έδρες προς 46 ε, αρκούν σε μια φυσιολογική χώρα για να έχει πλειοψηφία. Αλλά εδώ μιλούμε για κάτι ε, ουσιαώδες ως στρατηγική. Και όταν είναι διχοτομημένη η κοινωνία, είναι πραγματικά ανόητο να θεωρεί κάποιο ότι ο λαός της Μαλδαβίας είναι υπέρ της Ευρώπης. Δεν μ' αρέσει εμένα το αποτέλεσμα. Το λέω ειλικρινά. Αλλά αυτό είναι. Ακόμα και αν δεν μ' αρέσει, έτσι έχουν τα πράγματα και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ιστερία που έχει φιλορωσικό πληθυσμό, ο κόσμος εκεί δεν ψήφισε στις εκλογές, που είναι και μισό εκατομμύριο. Αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το θεωρούμε υποστήριξη στην ευρωπαϊκή ένταξη. Το λέω γιατί ξέρω ότι Μολδαβία εδώ και τέσσερα χρόνια ουδέποτε συνήντησα μια κατάσταση τελείως σαφή υπέρ της Ευρώπης αυτό που ξέρω εγώ αντικατοπτρίζεται στα παρόντα αποτελέσματα των εκλογών. Αν λαμβάνουμε επίσης υπόψη ότι μια τέτοια κρίσιμη ε, κατάσταση ε, συγκεντρώνει ένα 55,86% καταλαβαίνετε ποιος είναι ο ενθουσιασμός για την Ευρώπη και πάλι ε, αυτό, κορυδεύουμε τους εαυτούς μας με την Ουκρανία που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε πόσο φιλοευρωπαίοι είναι 52% είναι 52% Κοίταξε, μιλάω όσο μιλήσανε και άλλοι. Άμα δεν σας αρέσει τι να κάνουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να μην γελιόμαστε πάντως. Ε, η πραγματικότητα δεν είναι η ιδεολογία μας, είναι η αλήθεια. Mrs. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω στον πρόεδρο της αντιπροσωπείας, ίσως στον κύριο Κριστέ, αλλά μπορεί να σχολιάσει και ο κύριος Σόλτες. Ποια μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη βλέπετε τώρα να ε, υιοθετούνται μεταξύ Κίσιναου και Τυρασπόλ και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι για να εθαρρύνει αυτό το διάλογο για την ακαιρεότητα της χώρας. Και μετά πώς βλέπετε την κατάσταση του εμπορίου τώρα στη Μολδαβία. Ε, έχουμε τη συμφωνία σύνδεσης αφενός και αφετέρου την ε, ευρασιατική οικονομική κοινότητα με τη Ρωσία και το δικό της καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύεται ότι κάνει αρκετά για να βοηθήσει την Μολδαβία να διατηρήσει το εμπόριό της. Ευχαριστώ κύριε Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Το πρώτο μου σχόλιο αφορά τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Μπορούμε από τη μια να έχουμε φιλευρωπαϊκές δυνάμεις, ε, δηλαδή θέλουμε να τις φέρουμε αντιμέτωπες με άλλες δυνάμεις. Εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη αναζητούσε την ειρήνη και τώρα έχουμε θετήσει γλώσσα πολεμική. Από τη μια έχουμε φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και από την άλλη, δεν το λέμε, ε, φιλορωσικές δυνάμεις. Θυμίζω ότι η Ρωσία είναι μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρόλα αυτά ότι είναι τμήμα και της Ευρώπης γεωγραφικά και είμαστε εδώ σε ένα χάσμα, που, σε μια διαίρεση που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ιστορία, ούτε στον πολιτισμό μας, ούτε στην δημοκρατική μας νομιμοποίηση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερο, χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση. Ε, θα ήμασταν τόσο τρομαγμένοι αν ήταν η αμερικανική η χρηματοδότηση. Ε, κάποιος ε, είπε ότι δόθηκε ένα δισεκατομμύριο για την Ουκρανία από την Αμερική. Ρωτήστε τον κύριο Γιαννουκόβιτς πώς χρηματοδότησε την προεκλογική του εκστρατεία. Ας μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μια γλωσσία να είναι καλή χρηματοδότηση των Ηνωμένων ενώ η άλλη χρηματοδότηση να είναι κακή. Τρίτο σχόλιο. Τρίτο σχόλιο. Τρίτο σχόλιο. Τρίτο σχόλιο. Για τις προσωπικές επιθέσεις. Δεν σας είπα τίποτα, καθίστε κάτω σας Ναι, τρίτο σχόλιο. Για τις προσωπικές επιθέσεις. Είμαστε σε κράτος δικαίου. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Κύριε πρόεδρε, όχι. Προσωπικά, μου επιτέθηκαν και πρέπει να μου δώσετε το λόγο επί προσωπικού. Ο χρόνος σας τελείωσε. Τελείωσε ο χρόνος σας. Σας διακόπτω, διέκοψα και άλλους. Μπορώ να συνεχίσω. Ο κύριος Σόλτα. Please. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είπατε όλοι σας ότι στις εκλογές αυτό το οποίο καταδείχθηκε είναι ότι αποφάσισε η πλειοψηφία να ακολουθήσει ένα δρόμο που θα εγγυάται ε, τις πιο στενές σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία λόγω της γεωπολιτικής θέσης και της Ουκρανίας και άλλων ε, χωρών της Ανατολής. Και με τη Ρωσία. Εμείς έχουμε τονίσει και στο ψήφισμά μας ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως την γεωστρατηγική θέση της Ουκρανίας, λέει. Της οικονομική εμπορική κατάσταση στη Μολδαβία δεν είναι εξαιρετική και ούτε μπορεί να βελτιωθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι επίσης ε, γεγονός ότι η Μολδαβία από ενεργικής πλευράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από άλλες χώρες. Και φυσικά αυτό έχει επιπτώσεις και στη χώρα και στην κοινωνία. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Πάτρια, Πατρίδα και τη χρηματοδότησή του, πρέπει να σας πω ότι οι παρατηρητές των εκλογών επισημαίνουμε ότι με την απαγόρευση του κόμματος αυτού Γύρονται κάποια ερωτηματοκά, ιδίως σε ό,τι αφορά και το χρόνο που επελέγει για την απαγόρευση αυτού του κόμματος. Επιμείναμε επίσης ότι θα πρέπει να διασκεδαστεί κάθε αμφιβολία γύρω από την απαγόρευση αυτή. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ιδεολογική πολυμορφία, αυτό που επηρεάζει και την δημόσια κοινή γνώμη. Έλαμψη δια της απουσίας της ε, η πολυμορφία στον τύπο και στα μέσα επικοινωνίας, άρα δεν είναι αποτελεσματική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το ίδιο ισχύει και με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την υπερδυνιστερία και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διαδικασία αυτή πρέπει να σας πω ότι θα κρατήσει πολύ καιρό αυτή η διαδικασία. Το είδαμε και με τα ίδια μας τα μάτια. Υπάρχει έλεγχο στα σύνορα. Το θέμα είναι όμως, δεν είναι μόνο τα φυσικά σύνορα, αλλά τα... οι πώς μπορούν να αλλάξουν. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια πολύπλοκη και μακρά διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη που μίλησα ίσως κάπως σκληρά. Έχουμε κοντά μας και τους ε, φίλους μας της ε, Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής, της Bundestag. Θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της μέσης διδαξής μας της πολιτικής γειτονίας. Και βέβαια στη Μολδαβία σημειώνεται ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε δυνάμεις που θέλουν ένα κεντρικό σύστημα και σε αυτές που θέλουν μια ελεύθερη, φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτό ο αγώνα γίνεται και στη Γερμανία και σε πολλές άλλες χώρες και βλέπουμε ότι η χρήση των μέσων που κάνει η Ρωσία εκεί, η εμπορική περιορισμοί που επιβάλλει συστηματικά στη Μολδαβία η Μόσχα εδώ και δύο χρόνια και Ιδίω στον αγροτικό πληθυσμό εκεί με τα κόκκινα χρώματα που δείξατε και προσπαθεί να τους επηρεάσει να κινηθούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά και βλέπουμε να ενισχύεται το κόμμα εκείνο το οποίο χρηματοδοτήθηκε με τεράστια ποσά από τη Μόσχα. Ο Πούτιν ξεκίνησε μια τεράστια ε, εκστρατεία με αφήσει που τα μέσα της πόρη είναι άγνωστοι. Έθεσε ο κ. Μπιτικόφερ την ερώτηση πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην διαδικασία αυτή και να υποστηρίξουμε τα δίκαια της δημοκρατίας και τις δυνάμεις της δημοκρατίας που εν πάση περιπτώσει κέρδισαν τις εκλογές και έχουν και ξεκάθαρη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν νομιμοποίησή μας να το πράξουμε αυτό. Κέρδισαν λοιπόν τις εκλογές. Δεν θα ή να να αφήσουμε δηλαδή να επιπλέψουν οι άλλοι με τις παραλήψεις μας, αυτή την επιχειρηματολογία δεν μπορώ να τη δεχθώ ούτε από τον κύριο Νάτου, οποιοδήποτε κανέναν άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε ξεκάθαροι στις θέσεις μας αυτές. Πρόκειται μεν για μια έκτακτη περίπτωση μέσα στην πολιτική γειτονία, όχι όμως για μεμονωμένη περίπτωση. Και σε ό,τι αφορά την υπερδνηστερία, είτε πρόκειται για αυτήν, είτε πρόκειται για την Κρυμαία, είτε πρόκειται για την Απχαζία, είναι η ίδια κατάσταση. Παν να πετύχουν μέσα από την αποσταθεροποίηση κακή οικονομική απόδοση και τελικά να φορτώσουν την κακή οικονομική απόδοση των χωρών ε, στις δυτικές συμμαχίες. Όποιος δεν αντιλαμβάνει τη στρατηγική αυτή έχει ένα πρόβλημα συνολικότερα να κατανοήσει πού βρίσκεται η ελευθερία και η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Χαίρομαι που είναι παρόν και ο κύριος Πόστα. Από χθε είμαστε πανευτυχείς διότι λυπούμε πολύ Αλόης Πέτερλε η ομάδα μας κέρδισε και μπήκε στους πρώην τελικούς της Champions League. Μπορούμε λοιπόν να χαμογελούμε σήμερα. Γκίντερ, να σου δώσω το λόγο. Αν ναι, να έρθω πιο κοντά. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της Ευρωβουλής, πολύ ευχαρίστως ήλθαμε να σας δούμε σήμερα ως μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανικής Bundestag. Αυτά μέσα σε μια παράδοση που έχουμε που λέει ότι μια τουλάχιστον φορά το χρόνο διεξάγουμε μια εξωτερική επίσκεψη στις Βρυξέλλες έτσι ώστε να έρθουμε σε άμεση επαφή μαζί σας και βεβαίως και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μπορέσουμε να σας δούμε δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο. Εκτός από αυτό, ως μέλη βρισκόμαστε συχνά στις Βρυξέλλες, διότι, ως βουλευτές δηλαδή, διότι η Επιτροπή μας έχει στενή διασύνδεση και επιζητεί τη στενή αυτή διασύνδεση με τις και τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε άλλωστε και μοναδική επιτροπή όπου 15 οι Ευρωβουλευτές έχουν μόνιμη έδρα και σε εμά. Έρχονται δηλαδή όποτε θέλουν και μας παρακολουθούν. Μιλούμε για το θέμα αυτό σήμερα της ανατολικής πολιτικής γειτονίας που απασχολεί πάρα πολύ έντονα και την γερμανική Bundestag. Ως Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων το ζήτημα αυτό της ανατολικής γειτονίας και ιδίως τα γεγονότα στην Ουκρανία τα βάζουμε σχεδόν σε κάθε ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Με συμμετοχή σημαντικών επισκεπτών, είχαμε πρόσφατα τον Wolfgang Ischinger, επικεφαλής της ε, διάσκεψης ειρήνης και ασφάλειας του Μονάχου, πρόσφατα επίσης την καγκελάριο κυρία Μέρκελ. Είμαστε όμως και σε διαρκή επαφή με διάφορες ε, ομάδες προβληματισμού, think tank, και αυτά τα χρησιμοποιούμε και στις συζητήσεις μας για την εσωτερική πολιτική ακόμη και την εξωτερική πολιτική. Σας ευχαριστώ που σήμερα διαθέτετε το χρόνο για να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε τη συζήτηση αυτή από κοινού, να προχωρήσουμε δηλαδή σε μια συζήτηση μαζί σας, γιατί για μας η μοίρα των χωρών εκείνων που συμμετέχουν, που ήταν και εξακολουθούν να είναι στην ανατολική γειτονία, δεν μας αφήνει αδιάφορους. Αν κοιτάξουμε προς τα πίσω, ήταν έξι χώρες. Τρεις έχουν μείνει, Γεωργία, Ουκρανία και Μολδαβία. Και οι τρεις έχουν ένα κοινό στοιχείο. Και οι τρεις αυτές χώρες έχουν μια λεγόμενη παγωμένη σύγκρουση που έχει προκληθεί από τη Ρωσία βεβαίως και που εξακολουθεί να διατηρείται στη ζωή από τη Ρωσία είτε πρόκειται για τις συνομιλίες 5 2 στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας όπου τα πράγματα προχωρούν ελάχιστα στο θέμα της υπεδνηστερίας είτε πρόκειται για την Νότια Οσετία στην περίπτωση της Γεωργίας είτε πρόκειται για την νέα αυτή δημιουργηθήσα σύγκρουση την εισβολή δηλαδή στη Χερσόνησο Κρίμ, στην Κρυμαία και βεβαίως στα ανατολικά της Ουκρανίας, στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας. Βεβαίω, όλε αυτέ οι χώρε θέλουν ένα πράγμα. Να μοιραστούν μαζί μας αυτά που εμείς εδώ μοιραζόμαστε μεταξύ μας εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή τις ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της Ειρήνη, της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της δημιουργίας μιας βάσης κοινωνικής ασφάλειας και Έτσι αυτή η επιθετικότητα από πλευρά Ρωσία είναι μια επιθετικότητα και κατά των ευρωπαϊκών μας αξιών και γι' αυτό το λόγο αξίζουν οι χώρες αυτές την αλληλεγγύη μας. Έχουμε όμως και ένα σημαντικό συμφέρον στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει σταθερότητα. Γι' αυτό η Ανατολική Γειτονία είναι ας πούμε ένα υποσύνολο της εξωτερικής μας πολιτικής. Και εκτός από αυτό δεν πρέπει να λησμονούμε και τα γεγονότα στον βορρά της Αφρικής, όπου από την Αραβική Άνοιξη σε πολλές χώρες έχει πια φτάσει να μην πω ε, ε, αραβικός χειμώνας, τουλάχιστον αραβικό φθινόπωρο. Και εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε εμπλοκή. Και γι' αυτό αγαπητέ Έλμαρ Μπρόκ χαίρομαι πολύ που μας δέχεστε σήμερα ως φιλοξενουμένους σας και θα χαρώ πολύ να δω από κοντά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, μετά από την δική μου τοποθέτηση, αγαπητέ Έλμαρ, να ακούσαμε αγορητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, πάντοτε αναδύο από τα κόμματα. Αλλά ας ισχύσει χρόνος αγορεύσεως δύο λεπτών. Εσείς έτσι το έχετε εδώ. Εμείς είμαστε κάπως πιο γενναιόδοροι στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής. Δίνουμε τρία λεπτά. Όπως είδαμε όμως ότι είσαι αυστηρό στην τήρηση του χρόνου, δεχόμαστε να το πράξεις και για όλους. Ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που δίνετε για την διεξαγωγή αυτής της ζήτησης. Σου επιστρέφω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Δεν θα πω πολλά. Κάνω ωστόσο μια πρόταση πριν, έλθουν, πριν έρθουμε στις εκπροσώπους. Έχουμε την ε, κυρία Σαρλότε Σάμελιν της ομάδας υποστήριξης της Ουκρανίας πριν από συζήτηση με την κυρία Μογκερίνη μπορεί να μας πει σε λίγα λεπτά πώς οργανώνεται η διαδικασία αυτή τώρα από την ομάδα στήριξης αυτής στην ίδια την Ουκρανία. Πού είστε κυρία συνάδελφε. Σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε. Είναι μεγάλη τιμή για μας να παρευρισκόμαστε εδώ και να μιλήσουμε και ενώπιον των συναδέλφων από τη Γερμανική Βουλή. Αλλά θα μιλήσω αγγλικά ε, και να πω σύντομα αυτά που γνωρίζετε ότι έγιναν βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία στις 26 Οκτωβρίου και ήταν ένα σημαντικό βήμα στις προσδοκίες της Ουκρανίας να εδραιώσει τον εκδημοκρατισμό της όπως άλλωστε έχει δεσμευθεί ως χώρα. Στα πλαίσια αυτά και επί τη βάση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών θα πρέπει να αναζητηθεί στην Ουκρανία ευρύτερη συνένεση, εθνική συνένεση. Είναι πολύ θετικέ ε, οι προοπτικέ, η νέα ράντα, η νέα βουλή δηλαδή και η νέα κυβέρνηση έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσει να φέρουν ε, πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε συνεργαστεί και θα συνεργαστούμε στενά με την κυβέρνηση για την συνταγματική μεταρρύθμιση, την αποκέντρωση, ε, την ε, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνη, των διοκτικών αρχών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των κρατικών θεσμών. Με αυτές τώρα τις πολιτικές αλλαγές είναι ενώπιον νέας κατάστασης η Ουκρανία, νέα βουλή, νέο κυβερνητικό συνασπισμό που θα πρέπει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις και να βεβαιωθεί ότι θα εφαρμοστούν κιόλα. Είναι κρίσιμο αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Ε, σήμερα η κυβέρνηση έχει κληθεί στη Βουλή για να κάνει τις πραγματικές δηλώσεις για να εγκριθούν. Γενικά έχουμε την αίσθηση, που είναι πολύ γενική αίσθηση, ε, ότι είναι καλή η πρόοδος, καλό το πρόγραμμα, συνεχίζουν ε, την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Μεταρρυθμίσεων, συμφωνεί αυτό με το πρόγραμμα του κυβερνητικού συνασπισμού και με τις δεσμεύσεις της Ουκρανίας στα πλαίσια της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ε, το πρόγραμμα, το κυβερνητικό, ε, βασίζεται στις συστημικές αλλαγές όπως σας ανέφερα και στις πιο επίγουσες διαδικασίες για την σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας και του κράτους δικαίου. Τώρα θα πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία, δηλαδή και στην κυβέρνηση και στην Βουλή, το χρόνο και την ευκαιρία να εργαστούν. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις εξελίξεις ή την στάση τους. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά και από ποιες δομές. έχουμε νέο Υπουργικό Συμβούλιο ε, και οι Υπουργοί μπορούν να επιλέξουν τους υφυπουργούς τους οι οποίοι εργάζονται σε θέματα ευρωπαϊκής ένταξης. Η στρατηγική είναι σε ένα πλαίσιο 2015-2017, στρατηγική των μεταρρυθμίσεων εννοώ. Ελπίζουμε αρχές Ιανουαρίου το αργότερο να εγκριθεί Βεβαίως και αυτή η στρατηγική είναι πολύ σημαντική για το λαό της Ουκρανίας. Θα πρέπει η κυβέρνηση να είναι σαφής και με διαφάνεια να εξηγήσει και τους στόχους της. Συμπαρίσταται η διεθνής κοινότητα, αλλά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο το κυβερνητικό πρόγραμμα και η στρατηγική. Γιατί οι προγραμματικές δηλώσεις που κατατίθενται σήμερα στη Ράντα είναι πάρα πολύ γενικόλογες. Είναι ένα σύντομο κείμενο, έξι σελίδων. Εμείς θα θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα βήματα και πότε θα γίνουν αυτά. Πολλά θα εξαρτηθούν για την επιτυχία όλων αυτών ε, από την ε, προθυμία ε, της νέας ηγεσίας της χώρας να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή προσβλέπουν και στη δική μας υποστήριξη και ενθάρρυνση και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, στη δουλειά μας η λέξη κλειδί είναι το ownership, δηλαδή θα πρέπει να γίνει κτήμα τους αυτή η υπόθεση, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με συμβουλές, με βοήθεια, αλλά εκείνοι θα πρέπει να τα εσθενιστούν όλα αυτά, να τα υιοθετήσουν και να τα μεταφράσουν σε μια αξιόπιστη μεταρρυθμιστική στρατηγική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρεις γενικές παρατηρήσεις ε, για το θέμα που θα μας απασχολήσει. Θα αρχίσουμε σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επεξεργαζόμαστε την έκθεση για την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας. Θα έχω την τιμή, την ε, ευθύνη και τη χαρά να είμαι εισηγητής για αυτήν την έκθεση και νομίζω ότι έρχεται σε πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή, αν και η προηγούμενη έκθεση ήταν πριν από τρία χρόνια. Πριν τρία χρόνια αντιδράσαμε στις αλλαγές στην περιοχή, στο Νότο. Όπως επίσης είδαμε και την κρίση προς Ανατολάς. Τι έχουμε διαπιστώσει μετά από τρία χρόνια. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει πρέπει να μας γίνει, αν θέλετε, μάθημα. Δηλαδή, τέτοιες κρίσεις, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, φαίνεται ότι δεν ε, αποτελούν παρελθόν, θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο ρεαλιστές στον τρόπο με τον οποίο εκτιμούμε τέτοιες καταστάσεις που επαναλαμβάνω θα ξανασυμβούν. Και αυτό με βάση την εμπειρία που είχαμε πριν από τρία χρόνια ήμασταν ίσως υπερβολικά αισιόδοξοι σε σχέση με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα τελικά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν όλο το πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας. Η πολιτική αυτή πλέον θα πρέπει να έχει σαφείς μακροπρόθεσμους, συνεπείς στόχους και για τα δύο τη σκέλη. Κατέστη σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε εργαλεία πολιτικής μέσα για αυτή την πολιτική που θα συνάδουν με τους στόχους και αντίστροφα τα εργαλεία που θα στηρίζουν και την πολιτική μας ε, στην περιοχή αυτή. Στην αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας η απάντηση δόθηκε με βάση πιο πολύ τη δημοκρατία, ε, την ανάπτυξη και την συμμετοχή της κοινωνίας. Σωστή προσέγγιση, αλλά νομίζω θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσγειωμένοι και ρεαλιστές στην προσέγγιση μας στο μέλλον. Και θα πρέπει να μας απασχολούν περισσότερο ζητήματα όπως το εμπόριο, η ενέργεια, μετανάστευση, η ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, ο Μίχελ Στούπκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμεί χαιρόμαστε από πλευρά πολιτική ομάδα κοινοβουλευτική ομάδα τη ΕΝΤΕΟΥ Τσέσου για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε την επικαιρότητα τη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Και για μας είναι σημαντικό να μάθουμε πώς βλέπετε εσείς τις καταστάσεις και την ανάγκη να αναδιαμορφωθεί η ε, πολιτική γειτονία. Σύντομα θέλω να πω τα εξής. Πρώτον, ακόμα και αν ε, δεν ευθύνονται γι' αυτό οι εν λόγω ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Πολιτική γειτονία, όπως σχεδιάστηκε το 2009 και μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει στεφθεί ε, με τεράστια επιτυχία. Για διάφορους λόγους. Το ένα είναι η επιρροή της Ρωσίας, τα ίδια συμφέροντα της Ρωσίας σε πολλές από τις χώρες αυτές που ε, θα πρέπει να είναι μέλη της πολιτικής γειτονίας. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε πού είναι οι δικοί μας προσανατολισμοί και οι δικές μας ε, σκέψεις και που, κάναμε λάθη στις εκτιμήσεις μας. Να σας αναφέρω ένα σημείο που θεωρώ πολύ σημαντικό. Ανεξάρτητα από τη στάση της Ρωσίας που θεωρώ απολύτως απαράδεκτη στην Ουκρανία, θεωρώ όμως τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση άρον άρον να υπογράψει συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία, τη στιγμή που ούτε κατά διάνοια δεν ήταν πρόθυμη, έτοιμη ή σε θέση ε, να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία η Ουκρανία, για μένα είναι λάθος δρόμος. Ε, ε, το σημαντικό που προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που συζήτησε αυτόν τον καιρό είναι πώς μπορούμε στο μέλλον να προσανατολίσουμε καλύτερα την πολιτική γειτονίας χρειάζεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση και να ξέρουν ότι οι χώρες αυτές έχουν και ευθύνες και η πρόοδος και συνδέεται με την υποστήριξή μας. Δηλαδή υποστηρίζουμε όταν υπάρχει συγκεκριμένη πρόοδος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε με ενισχυμένο τρόπο προς τα εκεί, γιατί σε ό,τι αφορά τις χώρες αυτές της γειτονίας, δεν είναι χώρες που σε ένα ορατό μέλλον μπορούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν το αποκλείω, ε, γιατί δεν υπάρχουμε μόνο εμείς, υπάρχουν και επόμενες, υπερχόμενες γενιές. Αλλά και για τις χώρες αυτές πρέπει να γίνουν πρόοδοι σε θέματα συγκεκριμένα εμπορικά, τελωνιακά, συνεργασία, σε θέματα έρευνας κτλ. Ε, πλανάτε στο χώρο το μοντέλο της Νορβηγίας για άλλο λόγο. Η Νορβηγία είναι μια χώρα που είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι πλήρες μέλος. Ορίστε, θα μπορούσαμε μια τέτοια προοπτική να ανοιχθεί και για τις χώρες αυτές ως προσφορά με καλύτερες προϋποθέσεις και να ξέρουμε ξέρουν και εκείνοι τι θέλουμε, βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, από πλευράς του ΕΛΚ ε, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε διάλογο με τους ε, εθνικούς βουλευτές, τους συναδέλφους μας, να παραμένουμε σε επαφή για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την επίκαιρη κρίση της Ουκρανίας. Να είμαστε ενωμένοι και στην ανάλυση και στα μέτρα ε, και στα μηνύματα που στέλνουμε ότι αυτή η εισβολή για μας είναι απαράδεκτη και αναμένουμε να ε, ξαναβρει το δρόμο του διεθνούς δικαίου η Ρωσία. Τώρα, τι γίνεται συγκεκριμένα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους εμπειρογνώμονες αλλά και την πραγματογνωμοσύνη που έχουμε ε, να ε, είμαστε παρόντες σε σημεία κλειδιά της χώρας και εκείνοι που θέλουν ε, να κάνουν μεταρρυθμίσεις να έχουν τη βοήθειά μας. Προτεραιότητες ουσιαστικά δεν υπάρχουν γιατί είναι όλα κρίσιμα και πήγοντα αλλά εδώ υπάρχει ένας τομέας που κατεμένα προέχει είναι το σύνολο της εσωτερικής ασφαλείας στη χώρα. Δηλαδή και οι ακτιβιστές της πλατείας Μεϊντάν που τώρα έχουν μπει στη Βουλή είναι καμιά σαρανταριά ακτιβιστές που έχουν εκλεγεί ως βουλευτές από διάφορα κόμματα. Δεν έχει δοθεί συνέχεια σε αυτά τα γεγονότα. Ε, παραμένουν ακόμα οι παλιές δομές και πρέπει να τους βοηθήσουμε να ε, μεταρρυθμιστεί ε, η εσωτερική ασφάλεια για να το συνειδητοποιήσουν και οι άνθρωποι αυτοί γιατί έχουν την αίσθηση ότι είναι ακόμα υπαλλήλοι στα πράγματα. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ λοιπόν η συμφωνία αυτή σύνδεση που την αναβάλαμε για ένα χρόνο, θα πρέπει συγκεκριμένα να ασχοληθούμε εν μέρει και με τη Ρωσία να συνεννοηθούμε για τα τεχνικά ζητήματα έτσι ώστε να μπορούν αυτά να εφαρμόζονται καλύτερα. Αλλά δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι το σύνολο της συμφωνίας αυτής και η ουσία της θα πρέπει να εφαρμοστεί για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ σύνολη συμφωνία. Έχουμε καταργήσει τους δασμούς σε κάποιους τομείς για να βοηθήσουμε τη χώρα. Θα κάνουμε και άλλα βήματα πρόοδου στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που συζητούμε το θέμα εδώ όλοι μαζί και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές ότι αν εξετάσουμε την πολιτική γειτονίας προς, το, προς τα πίσω, στο παρελθόν δηλαδή, έχουμε σημειώσει και λάθη. Όχι μόνο σε χώρες που τους προσφέραμε την πολιτική γειτονία, αλλά όχι μόνο από τις ίδιες χώρες δηλαδή έγιναν σφάλματα, αλλά και από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. τους δίνουμε την ε, ελπίδα, την προσδοκία μιας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να τους θέλουμε πραγματικά. Έχει συμβεί αυτό. Γι' αυτό η πολιτική γειτονία πρέπει να είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη ότι δηλαδή θέλουμε γειτονικέ σχέσεις, θέλουμε συμφωνίες, θέλουμε συμφωνίες συνδέσεως που όμως δεν οδηγούν απαραίτητα και πάντως όχι σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια ενδεχόμενη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνάδελφός μου εδώ δίπλα μου, ο Άχιμ, θα μιλήσει σύντομα και για την πολιτική μας προς τη Μεσόγειο. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας απέχουν πολύ από του να πληρώνουν τα κριτήρια για την ένταξή τους. εξηγήσατε και πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα πολιτική γειτονίας. Θεωρώ ότι αν ξεκαθαριστεί περισσότερο ότι θα ωφεληθούν από την Σύμφωνια Συνδέσεως οι άνθρωποι, θα ωφεληθούν από την καθημερινότητα μιας γειτονικής σχέσης, τότε εν τέλει ίσως η ένταξη της χώρας τους στην Ένωση να μην τους φαίνεται πια και τόσο σημαντική. Όπως εξήγησε και η πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως πρέπει να φροντίσουμε την αποκατάσταση κράτους δικαίου. Αυτό δεν σημαίνει μονάχα καταπολέμηση της διαφθοράς. Σημαίνει επίσης και περιορισμό του συστήματος των ολιγαρχών που βλέπουμε πολύ συχνά σε χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Η κυρία Μογκερίνη θα αναλάβει τώρα την αρμοδιότητα για την πολιτική γειτονία. Αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα, διότι μαζί με τον Επίτροπο κύριο Χάν θα είναι συναρμόδια. Επίσης, θέλω να ζητήσω να ληφθεί περισσότερο υπόψη το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην πολιτική γειτονία από ό,τι έως τώρα. Γιατί και μέσα από τα επίπεδα αυτά μπορεί να επηρεαστεί η καθημερινή ζωή των ανθρώπων και να τους καταστούν πιο ορατά τα ωφέλη. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Σκάν. Σίγουρα η ιδέα για την περιφερειακή πολιτική γειτονία ε, στέφθηκε με επιτυχία. Έχει και κάποια ε, σφάλματα βέβαια και καλό είναι να αναθεωρούμε σε τακτά διαστήματα αυτά που κάνουμε. Για μένα το ιδανικό βέβαια θα ήταν να μην βλέπουμε μόνο ε, την περιφερειακή πολιτική γιατί σίγουρα έχουμε κάποιο κοινό παρονομαστή έτσι αλλά να δούμε και κατά χώρα συγκεκριμένα ποιες είναι οι ανάγκες, τι γίνεται. Παραδείγματο χάρη, Μεσόγειος, βλέπετε, Αίγυπτος από τη μια πλευρά ε, έχουμε τη συζήτηση για τη σταθερότητα. Βλέπετε όμως πόσο έχει πληγεί η δημοκρατική διαδικασία. Έχουμε κατάφαρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν συνέβαιναν ούτε επί περίοδου Μουμπάρα και έχουμε και διολίσθηση και μετακύληση όλων των κλιμάτων και στη γειτονική Λιβύη. Ε, τεράστιοι πόροι φυσικοί, πλούτος ε, ε, και έχουμε δει όλοι μας το ίσις και άλλες τέτοιες οργανώσεις ε, τι καταστροφή έχουν δημιουργήσει. Άρα σε κράτη που καταραίουν όπως η Λιβύη μπορεί οι καταστροφές να είναι ακόμη μεγαλύτερες. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει και η πτυχή της ασφάλειας σε αυτή την εξίσωση και να δούμε και ποια είναι τα ενδιαφέροντα ή συμφέροντά μας αλλά αναχώρα και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήδη τέθηκαν ορισμένα θέματα και επισημάνθηκαν σφάλματα. Το κύριο σφάλμα που αφορά την περίπτωση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας νομίζω είναι ότι μια χώρα η οποία κατά το μισό προσανατολίζεται προς την Ευρώπη και κατά το άλλο μισό προς τη Ρωσία τίθεται ξαφνικά ενώπιον μπροστά σε ένα δίλημα αυτή η κρίση προκλήθηκε και με την Συμφωνία Συνδέσεως που θα ψηφιζόταν πέρσι τον Νοέμβρη στην Βίλνιους, που θα υπογραφόταν μάλλον στην Βίλνιους πέρσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό δίδαγμα που πρέπει να συναγάγουμε. Και αυτό το δίδαγμα πρέπει να το εφαρμόσουμε και στην περίπτωση της Μολδαβίας. Λέχθηκε ακόμη ότι πρέπει να περιορίσουν τους ολιγάρχες στην, ε, Ουκρανία. Είχα την ευκαιρία φέτος να μεταβώ έξι φορές εκεί. Η εντύπωση που έχω, συναποκομίσει από εκεί, είναι ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα σε αυτό το ε, ολιγαρχικό σύστημα. Η Ουκρανία είναι μια χώρα όπου υπάρχουν, υπάρχει μια σδράκα υπερπλούσιων οικογενειών με εισοδήματα τα οποία απέκτησαν στις δεκαετίες του 90 και μετά και αυτοί υπαγορεύουν την πολιτική. Και δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε την Ουκρανία, θα πρέπει να συνδέσουμε την κύρωση της ε, Συμφωνίας Συνδέσεως και με αυτό το σύστημα των ολιγαρχών. Τώρα, για τη Συμφωνία Συνδέσεως, όπως είναι διατυπωμένη βρίσκω ότι είναι και αντίθετη με οποιαδήποτε έννοια κράτους δικαίου. Για τη Μολδαβία, πολύ σύντομα. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή μας μιλήσαμε και για τη Ρουμανία και ακούσαμε για απάτη, νοθεία για τις εκλογές, γιατί οι Ρουμάνοι που είναι κατεστημένοι στην Αλοδαπή δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν. Το ίδιο είδαμε και στη Μολδαβία, όπου πολλοί άνθρωποι που ήταν στη Ρωσία δεν επιτρεπόταν να ψηφίσουν. Και τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές απαγορεύτηκε ένα κόμμα το οποίο στα δημοψηφι... Ε, στις δημοσκοπήσεις έφτανε το 15%. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα να πω. Το κύριε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 12 χρόνια είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής και έχω διατελέσει εισηγητής και για τις αρχικά συνδυασμένες εκθέσεις, οπότε και είχαμε έναν και μόνο εισηγητή για την πολιτική γειτονία και το 2005 για την ανατολική γειτονία, για τις πτυχές ανατολικής γειτονίας, άρα νομίζω ότι είμαι αρκετά έμπειρος ε, τώρα το ένα μέγεθος για όλα, ε, Αζερμπαϊτζάν μέχρι Αλγερία, ε, είναι ένα μοντέλο που δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς εξελίχθηκαν οι πολιτικές συν το χρόνο. Και είδαμε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα και των ευρωπαϊκών χωρών ε, που μπορούν να, να γίνουν δυνητικά υποψήφιες χώρες δυνάμετα του 49. Και μιλάω για χώρες από την Ανατολική Ευρώπη, ε, υπάρχουν και άλλες όπως σε Μέση Ανατολή, ε, που φυσικά δεν εντάσσονται στο άρθρο 49. Έχουμε τη διαφάνεια, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, που πρέπει να προστατεύουν και έχουμε μια συνολική πολιτική που δεν ακολουθεί τις ομονωμένε πολιτικές. Πρέπει να πω βέβαια ότι είναι λυπηρό το ότι κατελήφθη με εξαπίνηση. Αν δείτε και τι έλεγε και εδώ και 10 χρόνια ο πρόεδρος Πούτιν, οι προθέσεις του ήταν από τότε ξεκάθαρες. Εμείς όμως ε, ε, δεν το καταλάβαμε. Ήθελε να δημιουργήσει ένα είδος ε, σφαίρας επιρροής τύπου Γιάλτας. Και βλέπουμε τώρα με τη λεγόμενη Ευρασιατική Οικονομική Ένωση που είναι το νέο του σχέδιο. Άρα το νέο του παράδειγμα ουσιαστικά παραβιάζει όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και δίκαιο από το Ελσίν και μετά. Και σίγουρα πρέπει να σεβαστεί την εδαφική ακαιρεότητα και την κυριαρχία της Γεωργίας, της Ουκρανίας, κάτι που δεν το πράττει και αυτό βέβαια είναι απαράδεκτο. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 28 κρατών μελών ε, για το θέμα της επιβολής κυρώσεων ε, στη Μόσχα. Η δική μας άποψη, η ομάδα ECR, θα ήθελε να καταγραφεί στα πρακτικά ότι εκφράζουμε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για την πολύ άτεγκτη ε, στάση της καγκελαρίου Μέρκελ και της Bundestag στο Βερολίνο που μίλησε υπέρ του κυριαρχικού δικαιώματος της Οκρανίας ε, να έχουν ε, τη δυνατότητα να ασκούν τις πολιτικές τους χωρίς να δέχονται εξωτερικές πιέσεις όπως βλέπουμε να γίνονται τώρα ε, με τον Ντόμπας και την Κρυμαία από τη Ρωσία. Αυτά λοιπόν και ευχαριστώ και να διαβεβάσετε τις ευχαριστίες μου στην Καγκελάριο. Uh, ευχαριστώ και εγώ να δούμε λίγο τη το μελλοντικό σχεδιασμό της στρατηγικής ανατολικής γειτονίας. Νομίζω πρέπει να αντικαταστήσουμε κάτι το καλύτερο. Που ωστόσο η ανατολική γειτονία, η πολιτική ανατολική γειτονία ήταν σημαντική για τα τελευταία 25 χρόνια. Επίσης δεν υπήρξε διαδικασία διεύρυνσης με το στόχο αυτό στο τέλος, με την ένταξη, την ένταξη των χωρών δηλαδή. Εάν μακροπρόθεσμα αλλάξουν ωστόσο οι χώρες αυτές θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρος στόχος και εφόσον εκφράσουν ελεύθερα δημοκρατικά τη βούληση για την ένταξη. Η στρατηγική ανατολική γειτονία πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι που να επιτρέπει την παραπέρα εξέλιξη. Η στρατηγική ανατολική γειτονία δεν μπορεί να υποκατασταθεί σε, αυτό το ενδεχόμενο ένταξη. Και βεβαίω αυτά πρέπει να τα αποφασίσει και το Συμβούλιο και όχι μόνο τα πράσινα κόμματα στην Ευρώπη. Ήδη από το 2004 έχουμε δει το Κρεμλίνο να προσπαθεί να φτιάξει ένα είδος state building, ας το πω έτσι, ή system building, για να κάνουμε τη σύγκριση στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο προσπαθεί να φτιάξει ένα σύστημα φασισμένο στα ρωσικά πρότυπα. Και απέτυχε. Τώρα είναι η σειρά μας να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να μεταρρυθμιστεί προς την κατεύθυνση του δικού μας συστήματος που βασίζεται σε αξίες. Και εδώ πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί η διαφθορά είναι αυτή που ανοίγει τις πόρτες στο Κρεμλίνο για να βάλει πόδι στη χώρα. Και πιο βραχυπρόθεσμα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Αν το Κρεμλίνο έρχεται να συμφωνήσει μαζί μας λόγω των κυρώσεων, πρώτα δεν πρέπει να σταματήσουμε να μιλούμε για την Κρυμαία. Δεύτερο, να δούμε να μην παρισφρήσει το Κρεμλίνο στην Ουκρανική πολιτική έτσι ώστε να την υπονομεύσει. Δεν συμφωνώ ότι έχουμε αδύναμη θέση απέναντι στην Μόσχα. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την διαφθορά να μην υπάρχουν πράκτορες πληρωμένοι από τη Μόσχα και στην Ουκρανική κοινωνία, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις δικές μας κοινωνίες. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους Γερμανούς συναδέλφους και προσβλέπουμε στη διαρκή συνεργασία μαζί σας. Έχω και μερικά θέματα που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κρίχμπαουμ και αν θέλει να απαντήσει. Μπορούμε να κατηγορούμε ορισμένες χώρες ε, της ε, γειτονίας ότι οι ολιγάρχες έχουν βάλει χέρι στην οικονομία τους. Αλλά τα λεφτά τους πού τα έχουν οι ολιγάρχες. Να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Σε ποιες χώρες έχουν καταθέσει αυτοί οι ολιγάρχες και σε ποιες τράπεζες. Να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη. Δεν είναι ρωσικές. Στη Δύση είναι τα περισσότερα ρωσικά χρήματα των ολιγαρχών. Να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά υπάρχουν και καλές ειδήσει και για την Ουκρανία και όντως, ε, σε αυτή τη χώρα βασίλευε η διαφθορά, αλλά τα πιο πρόσφατα νέα τι δείχνουν. Ότι δέχτηκε η Ουκρανία να δεχτεί τον κύριο σε μετά, τον πρώην επίτροπό μας στην Επίτροπη ε, Μπαρόσο, είναι ο ύπατος αρμοστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα κοιτάζει τι γίνεται στην Ουκρανία, τις επιχειρηματικές συμφωνίες και τις κρατικές προμήθειες. Αυτή είναι σπουδαία είδηση και μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι και καλό παράδειγμα αυτό. Και τέλος, η ενέργεια ε, θα πρέπει να παραμένει στρατηγικό στοιχείο οποιασδήποτε πολιτική στην Ευρώπη. Και θα παρακαλούσα τον κύριο Κρίχμπαουμ να μας πει αν είναι πρόθυμη η Γερμανία να προχωρήσεις και στην Ενεργειακή Ένωση, όχι Ενεργειακή Κοινότητα, κάτι παραπάνω. Και να ε, ρωτήσουμε και τις υποψήφιες χώρες, αν θέλουν, να τηρήσουν τα υπεσχημένα. Ε, γιατί έχουμε συμφωνίες ε, σύνθεσης, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διμερών συμφωνιών. Και χαίρομαι για τη γερμανική στάση για τη διατήρηση των κυρώσεων. Είναι το μοναδικό πραγματικό όπλο απέναντι σε οποιαδήποτε περαιτέρω εισβολή στην ε, Ουκρανία η επίθεση και θα πρέπει να διατηρούνται οι κυρώσεις μέχρι να ε, εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Μίνσκ και να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία. Και να υπάρχουν και, και οι συνοριοφύλακες, όχι μόνο αυτονομιστές και ε, ρωσικά στρατεύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω με τα σφάλματα που κάναμε και να αναφέρω δύο. Το πρώτο. Πολύ εύπιστα και με ε, ε, ε αθώο τρόπο και αφελή δεχτήκαμε τις επιδιώξεις της Ρωσίας που ε, ήθελε ένα είδος νέο δόγμα πρέσβευ να έχει μια ζώνη ουδέτερη επιρροή στη γειτονία της. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που περιγράψατε ότι ο πληθυσμός είναι μισός-μισός εκεί, ε, φίλο ρωσικός. Μαζί είχαμε πάει στην Οδυσσό και ήταν σχεδόν ρωσόφωνη η πόλη και μας είπανε οι ε, συνομιλητές μας ότι είναι υπερήφανοι Ουκρανοί Ρωσόφωνοι, δεν θέλουν καθόλου να ε, ενωθούν με τη Ρωσία. Το κέντρο μας είναι στο Κίεβο, είπανε, και η σοβιετική νοσταλγία ε, το κάποιων ηλικιωμένων είναι κάτι που αναφέρεται εκεί. Και επίσης υπάρχει ρωσική προπαγάνδα σε αυτές τις χώρες την οποία έχουμε υποτιμήσει εδώ και καιρό γιατί βάζουν σφήνα για να διχάσουν τον πληθυσμό με μοναδικό στόχο να τους αποσταθεροποιήσουν. Θα πρέπει αυτές τις απόπειρες αποσταθεροποίησης να τις αποκρούσουμε και πώς θα γίνει αυτό με σαφή προοπτική. Και για μένα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή προοπτική που είναι και η Συμφωνία Σύνδεσης και ε, μια προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν θα πρέπει να συγχέονται αυτά τα δύο. Συμπέρασμα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτοματισμός. Δεν επιτρέπεται ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική δεν σημαίνει ένταξη, αλλά να μην αποκλείεται και αυτή, γιατί ε, αυτό είναι κινητήρια δύναμη που χρειάζεται μια τέτοια όθηση στις χώρες αυτές για να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Από την αριστερά κυρία Λόζενγκ. Ε, ναι, εκπροσωπώ την ΚΟΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ό,τι φαίνεται επικρατεί συμφωνία ότι η πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να θεωρείται επιτυχημένο εγχείρημα σε ό,τι αφορά την Ουκρανία ή την Ανατολική γειτονία. Τα συμπεράσματα είναι απλά. Φταίει η Ρωσία, να πιέσουμε τη Ρωσία και τα πάντα θα διορθωθούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν να αναφερθώ κάπως γενικότερα στην πολιτική γειτονίας για να ε, μην ακολουθήσω απαραίτητο αυτό το μονοδιάστατο μονοπάτι. Ε, στην πολιτική γειτονία θα πρέπει οι επιχειρήσεις των χωρών αυτών χωρίς προστασία ε, να ανοίξουν τις αγορές τους και να ανταγωνιστούν δυτικέ επιχειρήσει σε μια ελεύθερη αγορά χωρί να είναι σε θέση. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα και για την Ουκρανία και τώρα που έρχεται να εφαρμόσει ε, την ε, Συμφωνία σύνδεση. Τα αποτελέσματα στα πλαίσια τώρα τη νότια γειτονία. νομίζω ότι έπρεπε να τα είχαμε προβλέψει. Για τις χώρες νότιας γειτονίας, ας πούμε, έχουν έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ 2006-2010 από 530 εκατομμύρια έφτασε στα 20,4 δισεκατομμύρια το έλλειμμά τους. Και αυτό ήταν ε, κάτι το οποίο πυροδότησε και την Αραβική Άνοιξη. Δεν φταίει για όλα η Ρωσία σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Ήδη υπάρχουν προβλήματα από την εφαρμογή ε, των όσων ζητάει η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ε, φτωχοποιεί το λαό της χώρας σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις. Και χωρίς την επιρροή της Ρωσίας, να το πω λίγο κοινικά, αυτό ε, που εκτρέπει μια χώρα και τη διχάζει είναι η φτωχοποίηση του λαού της. Αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου εδώ μέσα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουμε την πορεία μας όπως την έχουμε χαράξει και στην νότια γειτονία και παντού. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας οπωσδήποτε. Μπάρχμαν, Σοσιαλδημοκράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε με τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Εγώ ασχολούμαι τώρα περισσότερο με την νότια γειτονία, με τις χώρες της Βορειοαφρικής δηλαδή και από τη Γερμανία είμαι και μέλος της Κοινοβουλευτικής συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και συμμετέχω σε πάρα πολύ χρήσιμες όσο και ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις που ασχολούνται με την πολιτική, τον πολιτισμό, την οικονομία, τις γυναίκες, την ενέργεια, το περιβάλλον με τρόπο πάρα πολύ εντατικό. Σημειώνω αυτό που είπε ο πρόεδρος ότι από την Αραβική Άνοιξη έχουμε φτάσει σε ένα αραβικό φιδινόπορο. Αλλά υπάρχουν και θετικές εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική. Βλέπε ε, κυρίως την Τινησία, όπου διεξήχθησαν εκλογές και έδειξαν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος που μπορεί κανείς να ακολουθήσει για να προχωρήσουμε κάπως. Γι' αυτό θα ήμουν πάρα πολύ υπέρ και εγώ της πρότασης η νότια πολιτική γειτονίας να γίνεται περισσότερο αντιληπτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δίνει περισσότερη προσοχή. Υπάρχει η λεγόμενη διαδικασία της Βαρκελόνης, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει δρομολογηθεί και ακολουθεί την πορεία της. Äh, και στη Μεσόγειο έχουμε πολλά μεταναστευτικά ε, ε, ρεύματα, ε, κάτι που κάνει το θέμα πολύ πιο επίκαιρο. Και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα θέμα που θα πρέπει και αξίζει να το σκεφτούμε και να το συζητούμε, γιατί αξίζει την προσοχή μας. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή μας ε, που διοργάνωσε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ε, γενικά οι ε, ανταλλαγέ απόψεων μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι πολύ θετικό και θέλω εδώ να ευχαριστήσω που οι Γερμανοί ομολογοί μας συμφώνησαν με τη διατήρηση του καθεστώτος κυρώσεων. Αν δεν είχε γίνει αυτό δεν θα ήταν καλή εξέλιξη. Τώρα έρχομαι στο γενικό ζήτημα ανατολική γειτονία και γενικότερα πολιτική γειτονία. Βλέπουμε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι. Οι παλέ πολιτικέ μπορούμε να ε, πούμε τι απόψει μα κάτω πόσο ήταν επιτυχημένε ή όχι, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να συνεχιστούν ε, όπω μέχρι τώρα. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι και έχουμε μπροστά μα μια επιλογή. Είτε να πούμε ότι τελικά θέλουμε μια ε, ένα μακροπρόθεσμο σύστημα ή καθεστώς που θα οδηγήσει ε, στο απότερο ή πολύ απότερο μέλλον σε ένταξη ή θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική δέσμη πολιτικών ανάλογα με τις περιοχές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε και προεδοπέ για αυτό είναι ε, άλλο να λέμε και άλλο να κάνουμε. Δηλαδή, άπαξ και ληφθεί μια σαφής απόφαση και όταν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο θα σας πω εγώ ποια είναι δική μου προσωπική άποψη, ε, μετά θα δούμε. Αλλά πρέπει να είναι σαφής η έκβαση των πολιτικών γειτονία. Τώρα, ε, πιο πολύ για την νότια γειτονία, αλλά ισχύει και για την ανατολική. Ναι, more for more είναι μια στρατηγική που μπορεί να λειτουργήσει, αλλά υπάρχει και το less for less. Δηλαδή, τι κάνουμε όταν η άλλη πλευρά δεν ε, αποδίδει σε σχέση με αυτά τα οποία τις έχουμε ζητήσει. Μειώνουμε και εμείς αυτά που προσφέρουμε ή όχι. Πρέπει να προσέξουμε να μην κατεβούμε σε να μην μπούμε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Επίσης, έχουμε κάποιες τακτικές κινήσεις της Ρωσίας. Δεν θα πρέπει κανείς ε, να ε, τεθεί όμοιρος αυτών των εξελίξεων. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε από τη Ρωσία και να προσπαθήσουμε να το επιβάλλουμε. Ευχαριστώ. Εγώ έχω το λόγο, όχι, κύριος Καστάλντο. Σα ε, eh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς πρέπει να παρατηρήσω ότι η Ostpolitik έχει ε, αρκετή ε, έμφαση, όχι η Ζουντ πολιτικ. Δεν κάνουμε πολλά για τον Νότο όσο για την Ανατολή δηλαδή. Θέλω να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας από τη Γερμανική Βουλή. Πόσο όμως ε, συζητείται ο Νότος εδώ. Κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν ε, για το καθεστώς ε, κατάρρευσης κρατών όπως η Λιβύη και τα λοιπά. Εγώ νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Έχει ήδη καταρρεύσει η Λιβύη. Έχουμε εκπαίδευση τζιχαντιστών σε στρατόπεδα στην Ανατολική Λιβύη. Δεν υπάρχει ασφάλεια συνόρων. Υπάρχει συνεργασία πολλών ομάδων με την Αλκάιντα ε, στο Μαγκρέπ που έχουν πει αυτές οι ομάδες ε, ότι θα ε, συνεργαστούν με το χαλίφι του Ισλαμικού κράτους και θα συνεχίσουν μαζί του τον αγώνα. Στην Τινισέ είχαμε μια καλή εξέλιξη και σίγουρα πρέπει να στηρίξουμε την αναδυόμενη δημοκρατία εκεί και να βοηθήσουμε σίγουρα με τις εξελίξεις ε, μήπως θα έπρεπε η τίνηση να είναι ομόλογη, μάλλον οι συνομιλητέ μας με όλη ε, την περιοχή τελικά, ε, να είναι διαμεσολαβητές. Επίσης, ε, στο έτος του Μάρε Νόστρουμ, ...144 εκατομμύρια θα δώσουμε για αυτό το μέτρο, για αυτή την πολιτική... ...ενώ πεθαίνει κόσμο κόσμος στη Μεσόγειο ακόμη είναι πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και τις φυσικές καταστροφές στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και δεν ε, θα πρέπει μόνο η Ιταλία να ε, δέχεται όλο αυτό το φορτίο και το βάρος των μεταναστών. Έχουμε και τα προβλήματα με Ισπανία, Ελλάδα, τι γίνεται στη Μεσόγειο γενικά. Χρειάζεται βοήθεια όλων και οι Γερμανοί πρέπει να μας βοηθήσουν και αυτοί για να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε για την εξέβριση πολιτικών λύσεων ώστε να τις στηρίξουν αυτές βέβαια όλοι, όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Καλνιέτε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τους Γερμανούς συναδέλφους της Bundestag και να συγχαρώ επίσης την Τσέντεου για την επανεκλογή της Άγγελα Μέρκελ ε, ως Προέδρου του κόμματος. Και μπορούμε να συγχαρούμε και την Ευρώπη για την επανεκλογή της κυρίας Μέρκελ. Όπως γνωρίζετε τέλη Μαΐου στη Ρήγα θα έχουμε μία σύνοδο κορυφής ε, για την Ανατολική Γειτονία. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι προς το παρόν η Ανατολική Γειτονία είναι το μόνο πλαίσιο που έχουμε για την άσκηση πολιτικής γειτονίας με πολλές γειτονικές μας χώρες. Ενώ Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Λευκορωσία γιατί οι άλλες τρεις, Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία, ήδη έχουν υπογράψει συμφωνίες ε, σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι φιλοδοξία έχει λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής στη Ρήγα. Θέλουμε να δούμε πώς θα διαφυλάξουμε αυτή την πολιτική και για να γίνει αυτό θα πρέπει ίσως να την αναθεωρήσουμε και να την επανεξετάσουμε για να είναι πιο ευέλικτη στην ε, εφαρμογή της και να υπάρχει και περισσότερο οικονομική διάσταση στην πολιτική αυτή. Είναι πραγματική στρατηγική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση η πολιτική αυτή η γειτονία, διότι μπορούμε σε αυτόν τον τομέα να ανταγωνιστούμε με τη Ρωσία για να κερδίσουμε και επιρροή αλλά και ε, τον κόσμο, τον λαό των χωρών αυτό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να δούμε πώς θα δίνουμε περισσότερους πόρους και να ενημερώνουμε περισσότερο για την Ευρώπη στις χώρες αυτές και τις δικές μας αξίες. Ευχαριστώ. Mr. Zarazin. Ah, by having the occasion having a second round, I just wanted to say something. Okay, επειδή έχουμε το χρόνο να πούμε, να πω κάτι που δεν έχει υποθεί μέχρι τώρα. Νομίζω ότι εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταλάβετε και να προωθήσετε μια πιο ε, ενοποιημένη, ε, ένα πιο ενοποιημένο θεματολόγιο και εντός των θεσμικών οργάνων και μεταξύ ε, θεσμικών οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω θα έχουμε μία συνεδρίαση χρηματοδοτών σε αρχές του επόμενου έτους που θα πρέπει πιστεύω να συνδεθεί με διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, καταπολέμηση διαφθοράς και άλλα θέματα και για την Ουκρανία και για άλλες χώρες. Ε, μελλοντικά θα δούμε και άλλες εταιρικές σχέσεις και θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές ε, να είναι εταίρος μας, ε, αρρωγός των προσπαθειών μας. Σίγουρα θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ενωπημένη προσέγγιση όλων των θεσμικών οργάνων, παραλαμβάνω και σε σχέση και με τα κράτη-μέλη για την Ουκρανία και άλλες χώρες και νομίζω ότι αυτό είναι το καθήκον μας για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. να μην γνωρίζει η δεξιά τύπη η αριστερά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να έχουμε μια ενοποιημένη στρατηγική. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Chairman. Ο ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχά ε, χαιρετίζω την διοργάνωση αυτή τη συνάντηση που έρχεται σε πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή. Οπότε και πρέπει να ξανασκεφτούμε πολλά από τα έργα και σχέδια που είχαμε για τι ε, εξωτερικέ μα δράσει μεταξύ ε, αυτών και την ανατολική ή νότια εταιρική σχέση. Κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχει δραματική ανάγκη για καλύτερη συνεργασία και συντονισμό θεσμικής φύσεως και με τα περιφερειακά κοινοβούλια. Έχοντας υπόψη πόσο πολύ πλοκός είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής. Άπαξ και πρέπει να εγκριθούν οι στρατηγικές. Δεύτερον, εξίσου σημαντικό είναι να δούμε ότι αν η Ευρώπη θέλει να διαδραματίσει τον παγκόσμιο ρόλο της και να αξιοποιήσει το δυναμικό της, μποστινάρου λέγομαι. Πρέπει πρώτα-πρώτα να χαράξουμε μια στρατηγική η οποία θα προσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμό και όχι κάποια κράτη-μέλη μεμονωμένα. Επίσης, πρέπει να υπάρξει ένα σαφές αυτό καλύτερο σε συντονισμός και συσχέτιση της εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και των, διεθνών ε, συμφωνιών εμπορίου και ενέργειας. Η Φεντερίκα, που είναι η πατεκπρόσωπος τώρα, έχει και την αρμοδιότητα να είναι η συντονίστρια. Θα συμμετέχουν και άλλοι επίτροποι, αλλά εξίσου σημαντικό είναι και τα εθνικά κοινόβουλια να συμμετέχουν. Τέλος, αφού βιώσαμε την κρίση Ουκρανίας-Ρωσίας, πρέπει να δούμε τι αμυντικές δυνατότητες έχουμε, τι αμυντική απάντηση μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τιμές παραδείγματος χάρη όπως διαμορφώνονται και τι αμυντικές δυνατότητε έχουμε συμπληρωματικά ως προς το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ. Πάει η περίοδος ε, των ψευδεστήσεων ε, και της αυταπάτης. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση real politik. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι πραγματικά πρωταγωνιστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ και εγώ Ευχαρίστω δεύτερο λόγο. ιδίως για να ευχαριστήσω εγκαρδίως και εσάς κύριε Πρόεδρε και τον δικό μας Πρόεδρο που διεξάγεται αυτές τις κοινέ συνεδριάσεις. Είναι απαραίτητο, ιδίως στους τωρινούς καιρούς, να μιλούμε με μια φωνή και οι θέσεις που εκφράζουμε στην πολιτική γειτονία να είναι μάλιστα και συντονισμένες διακομματικά. Ένα παράδειγμα, του πρόσφατου παρελθόντος που με ανησυχεί ιδιαίτερα. Μιλήσαμε για τις ρουμανικές προεδρικές εκλογές και εγώ πραγματικά ανατρίχιασα όταν διαπίστωσα ότι ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργό εξέφρασε θέσεις με, για την επανένωση του ρουμανικού λαού με τον Μολδαβικό και χρειάστηκαν τρεις μέρες να περάσουν για να τον μαζέψουν. Με αγανάκτησε επίσης και ότι ο δικός μας αναπληρωτής καγκελάριος Σίγμαρ Γκάμπριελ συμφώνησε. Αυτά είναι δηλητήριο μέσα στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Και προκαλούν τα αμυντικά αντανακλαστικά της ρωσικής κοινοπολιτείας. Είναι απαραίτητο να σταματήσουν αυτά. Ευχαριστώ που φέρατε ε, και τον κύριο Γκάμπριελ στο παιχνίδι όπως προηγουμένως κάποιος την κυρία Μέρκελ. Ο κύριος Κριστέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω χρειάζεται μια ισορροπία σε αυτή την επαναδιατύπωση της πολιτικής γειτονίας ανάμεσα στην ανατολική διάστασή της και στην νότια διάστασή της προς τη Μεσόγειο. Είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή προοπτική να, να, να λεχθεί μάλλον ότι η ευρωπαϊκή προοπτική υπάρχει μοναχά τώρα για τους ανατολικούς εταίρους. Τώρα εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Υπάρχει μια στρατηγική, υπάρχουν κάποιες γραμμές ε, σε σχέση με τη διάσκεψη κορυφής της Ρήγα τον επόμενο Μάη. Έχουμε εκεί να αναμένουμε θα αναμένουμε μάλλον θα πρέπει να αναμένουμε εκεί αίτηση εντάξεως σε χώρας. Das Δεν το άκουσα. Θέλω να επανέλθω σε μια σκέψη που άκουσα πριν για την κρίση με την Ουκρανία και με τη ρωσική στάση. Μέσα από όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις χώρες της νότιας γειτονίας. Η κατάσταση εκεί είναι εκρηκτική. Παράδειγμα, που δεν έχει ακουστεί στην συζήτηση που γίνεται δημόσια για την Αίγυπτο. Υπάρχουν διαρκώς ένοπλες επιθέσεις, γίνονται διαρκώς ένοπλες επιθέσεις των μουσουλμάνων αδελφών για να αποσταθροποιηθεί το σύστημα. Γίνονται απαγωγές, φόνοι και μάλιστα και μεγάλων αριθμών που δεν αναφέρονται εδώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προ λίγων ημερών επισκέφθηκα το κοπτικό κέντρο. Μπροστά βρίσκονται δύο τεθωρακισμένα και σταθμοί με πολυβόλα. Φανταστείτε τώρα τι κατάσταση. Το τελευταίο καιρό έχουν κάψει 78 εκκλησίες. Αυτό δείχνει εδώ πόσο βάναυσα προχωρούν, πόσο βάναυσα δρούν οι φονταμενταλιστές εκεί, ιδίω οι μουσουλμάνοι αδελφοί. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ρίξουν την κυβέρνηση. Γι' αυτό η παράκλησή μου προς εσάς είναι να μην παραλείψουμε να δράσουμε. Δηλαδή να λάβουμε παρόμοια μέτρα και εκεί όπως αυτά που συζητήθηκαν προηγουμένως για τη Μολδαβία. από εμάς, εμείς μάλλον χρειάζεται να στηρίξουμε αυτή τη διαδικασία εκδημοκρατισμού που προχωρεί πάρα πολύ αργά, είναι γεγονός. Και όχι βέβαια με στήριξη του στρατιωτικού καθεστώτος, αλλά να λάβουμε τα άλλα μέτρα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ja, zunächst